Dear colleagues, good morning. Since we are limited in time, let us... Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ας ξεκινήσουμε ε, το σημείο υπερθμών 1, έγκριση της σημερινή διάταξης. Και θέλω να σας ενημερώσω ε, τα 7, 8, το 60 και το 35 να ε, αναβληθούν. Το 9 μετά το 29 ε, τα 30 και 31 μετά το 24 και το 40 να εξεταστεί μετά το 14. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, ως εκ τούτου ε, θεωρώ ότι όλα αυτά εγκρίθηκαν. Το υπαριθμόν 2 ανακοινώσεις του Προέδρου Πρώτα απ' όλα ε, να μην ξεχάσετε να πάρετε τις ε, κάρτες σας ε, για αύριο το πρωί και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη συνάντηση θα την ολοκληρώσουμε σε 9 και 50 και θα σας καλέσω να έρθετε μαζί μου για να τιμήσουμε τα θύματα του 2016 της τρομοκρατικής επίθεσης της Βρυξέλλες. Αυτή η τελετή θα λάβει χώρα στον τρίτο όροφο ε, μπροστά στην Ολομέλεια. Ε, ε, Συνεχίζουμε λοιπόν με την κανονική μας συνεδρίαση με την Επιτροπή ΙΜΚΟ, την κοινή. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ντίτα Χαράντσοβα, αντιπρόεδρο της ΙΜΚΟ και τα μέλη της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ. Και θα ήθελα <clears throat> να σας ανακοινώσω ότι ο στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες. Έχουμε 988 τροπολογίες. Βεβαίως δεν έχουμε χρόνο να τις συζητήσουμε όλες ε, λεπτομερώς, αλλά ε, περιπτώσει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην την κυρία Χαράτσοβα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω ε, σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για σας, γιατί για πρώτη φορά ε, θα έχουμε στην ιστορία του Κοινοβουλίου δύο ε, συναντήσεις των δύο επιτροπών μας και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στους ε, δύο συνεισηγητές μας και θα θέλαμε να ακούσουμε τα δικά τους τα σχόλια για τις ε, τροπολογίες που προτείνονται όπως επίσης και για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Κύριος Βος, Αξιλ Βος, είναι ο πρώτος συγητής. Παρακαλώ κύριε Βος, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Ε, χαιρετίζω κυρίως ε, την κυρία Γκέπχα, την ε, συνεισηγήτριά μου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής. Έχουμε, όπως ακούστηκε, 988 τροπολογίες. Αυτές τις τροπολογίες τις έχουμε ταξινομήσει σε διάφορες κατηγορίες και χτες το βράδυ συζητήσαμε, παραδείγματο χάρη, για το πρόβλημα του αποκαλούμενου embedded software. Ε, δηλαδή το πώς είναι δυνατόν ε, κατά κάποιον τρόπο να το ρυθμίσουμε αυτό το λογισμικό και καταλήξαμε στα γνωστά μας αποτελέσματα. Θέλουμε να βρούμε μια καλή προσέγγιση. Μια προσέγγιση η οποία ε, δεν θα, δίνει μόνο, δεν θα προσφέρει μόνο νομική σαφήνεια, αλλά θα δίνει και τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ε, νιώθει προστατευμένος ως προς τα δικαιώματά του. Και νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά θεμάτων που πρέπει να ρυθμιστούν με βάση βέβαια αυτές τις ε, τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί. Η κυρία Γκέπχαρ, θα τα δείξει όλα αυτά τα θέματα. Εγώ έτσι ε, απλά θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε ε, τελικά ε, ο τομέας εφαρμογής και αυτή η έννοια των δεδομένων ως ε, ανταπόκριση, κατά πόσον αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Θα πρέπει όμως ε, να συζητήσουμε και για την πλήρη εναρμόνιση αυτής της πρότασης και όσον αφορά την πλήρη εναρμόνιση, ε, με αυτήν σχετίζονται διάφορα θέματα ε, που έχουν σχέση με την ιεράρχηση των νομικών συνεπειών και με την δυνατότητα ενδεχομένως να καταγγελθούν οι συμβάσεις. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι το βάρος της απόδειξης και ε, οι ημερομηνίε αδειοδότηση. και αυτά τα δύο μα ενδιαφέρουν και υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά. Εμεί ω ΕΛΚ αυτό το οποίο κάναμε και το πώς ακριβώς τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά είναι ότι το θέμα που αποκαλείται Any Other Data, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον τομέα εφαρμογής, εκεί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτά τα any other data κάποιε άλλε μορφή δεδομένα, γιατί θα πρέπει αυτά να τα συμπεριλάβουμε. Γιατί κατ' ουσίαν ε, κίνδυνο βλέπουμε μόνο σε δεδομένα που έχουν σχέση με ανθρώπους, με άτομα, όχι οποιασδήποτε άλλη μορφή δεδομένα. Για το λόγο αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν κατανοώ γιατί πρέπει να τα συμπεριλάβουμε και τα άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα είναι, αυτό θα είναι αντικείμενο των ε, συζητήσεων. Πέρα από αυτό έχουμε ως ε, ΕΛΚ και τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις, τις οποίες τις ε, διαγράψαμε, γιατί δεν κατανοούμε γιατί εκεί πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν ήδη ε, για 24 μήνες ή για 5 χρόνια και δεν ξέρω ε, κατά πόσον θα πρέπει να διακόψουμε την ελευθερία σύναψης ε, σύμβασης με κάποιο δικαίωμα του καταναλωτή που αφορά στο μέλλον και που κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται καν να υπάρχει εναρμόνιση. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι αντικείμενο διαφορετικών απόψεων. Εγώ θεωρώ όπως σας είπα ότι το το είναι ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για την πλήρη εναρμόνιση, για τα δικαιώματα χορήγησης, ε, ε, τι επίπεδο επιθυμούμε ως προς αυτό και αυτό που ενδιαφέρει είναι επίσης και η αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Όλα αυτά ε, θα πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά. Όσον αφορά τώρα την αποζημίωση, ε, κατ' ουσίαν θα πρέπει να σκεφτούμε το αν όντως χρειαζόμαστε εναρμόνιση, διότι στα κράτη-μέλη Υπάρχει ήδη ένας κανονισμός περί αποζημίωσης, ο οποίος ε, κανονισμός ε, ρυθμίζεται και με βάση ή βασίζεται και στην παράδοση που ισχύει στο κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, για μένα δεν είναι απόλυτα κατανοητό το γιατί θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με αυτήν την πρόταση. Όσον αφορά τώρα τα δεδομένα και τις ε, νομικές συνέπειες, ε, μέχρι τώρα έχουμε ακολουθήσει ένα πολύ καλό δρόμο. Λέμε δηλαδή δεδομένα που έχουν σχέση με συγκεκριμένα άτομα και τα σχετικά συμβασιακά πρότυπα καλύπτονται από το βασικό κανονισμό περί προστασίας δεδομένων και δεν πρέπει και δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα επιπρόσθετο καθεστώς με επικαλύψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχατ, συνεισηγήτρια από την ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Axel ε, για την ε, μέχρι τώρα καλή συνεργασία, παρότι σε ορισμένα θέματα ε, δίστανται πλήρως οι απόψεις μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα αναζητήσουμε κάποιες λύσεις από κοινού με τους συναδέλφους μας, τους σκιώδης ηγητές. Βεβαίως, ο δρόμος αυτός ε, θα είναι ε, πόντινος και πίπονος. Το διαπιστώσαμε αυτό χθε στις συζητήσεις. Εμείς ε, καταλήξαμε σε μια συμβαστική πρόταση. Δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσουν και οι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό το ότι μεριμνήσαμε να υπάρχει σαφήνεια. Το, ποια θα πρέπει να είναι η ορισμός ε, του digital content ε, σε σχέση με την ε, οδηγία περί του δικαίου πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός, να ξέρουμε τι εντάσσεται που και όλοι μας είπαμε, θα το πω έτσι απλά, ό,τι έχει σχέση να κάνει με δεδομένα ε, είναι αντικείμενο ε, της οδηγίας περί ψηφιακού περιεχομένου. Και μόνο όπου πρόκειται ε, για προϊόντα τα οποία δεν είναι ψηφιακού περιεχομένου, μόνο αυτά θα πρέπει εντάσσονται σε κάποια άλλη οδηγία. Επ' αυτού υπάρχει ομοφωνία στο Κοινοβούλιο και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ καλό, παρότι βέβαια προσπαθούμε να το ορίσουμε το ποιος ακριβώς πρέπει να είναι ορισμός, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μια μια καλή λύση. Όσον αφορά τώρα στο θέμα των, όπως αναφέρει και προηγουμένως, any other data, εγώ ε, διαφωνώ με τον κύριο Φως. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή θα πρέπει αυτό να το αφήσουμε στην οδηγία και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, ε, στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί. Δηλαδή, ε, υπάρχει διαχωρισμός ε, με το ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα, ποια δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι δύσκολο να βρεθεί βέβαια τέτοιου είδους ορισμός. Και κατά δεύτερον υπάρχουν ε, ορισμοί οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς και για το λόγο αυτό, για να μην υπάρχουν ε, κενά, θα πρέπει τα άλλη μορφή δεδομένα, τα any other data, να τα αφήσουμε και να πούμε ότι δεδομένα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με συγκεκριμένα άτομα, ότι αυτά καταρχήν αφήνονται κατά μέρο. Ε, ίσως αυτή να είναι μια συμβαστική πρόταση, αλλά τα δεδομένα κάποια άλλη μορφή δεν θα πρέπει να τα διαγράψουμε πλήρω. Τώρα, όσον αφορά τις ε, διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, ε, θα πρέπει να πούμε ότι ο στόχος μας δεν είναι να αλλάξουμε το βασικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, αλλά να ε, ξεκαθαρίσουμε ότι οφείλουν να τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές και αν δεν τηρούνται τότε αυτό οδηγεί στο να καταγγέλλεται η σύμβαση. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές διότι δεν αρκεί να έχουμε ένα βασικό κανονισμό ε, τον οποίο να μπορεί κανείς να επικαλείται αλλά σε τελική ανάλυση αν δεν ε, τηρείται ο κανονισμός αυτός ε, τότε να μην υπάρχουν διατάξεις για να εφαρμόζει το κανονισμό. και γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι απόλυτα σαφής οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα κατά τα άλλα και εγώ θεωρώ ότι ε, το θέμα της εναρμόνισης ε, πρέπει να το ορίσουμε στο τέλος. Ε, νομίζω ότι έχω πει επανειλημμένα αυτό, διότι κατά την άποψή μου αυτό εξαρτάται από το πώς ακριβώς ορίζεται η προστασία δεδομένων στην οδηγία. Αν προβλέπετε ουσιαστική και έντονη προστασία δεδομένων, τότε και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και τάσομαι υπέρ της πλήρους εναρμόνισης. Αν όμως η προστασία δεδομένων είναι περιορισμένη, τότε εγώ ε, προτιμώ τα κράτη-μέλη να δίνανται να ε, διατηρήσουν ή να προχωρήσουν προς ουσιαστικότερη προστασία δεδομένων. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το γνωρίζουμε προς το τέλος, όταν δηλαδή ε, θα γνωρίζουμε πώς ακριβώς ορίζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος, τα remedies. Σήμερα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι καταρχήν θα δω τις προτάσεις του ΕΛΚ και των φιλευθέρων, αν ε, περάσουν αυτές οι προτάσεις, εγώ δεν δέχομαι την πλήρη εναρμόνιση. Αν όμως οι πολιτικές ομάδες θέλουν να προχωρήσουμε, τότε και εγώ μπορώ να αναθεωρήσω λιγάκι την ε, πρότασή μου. Και γι' αυτό έχω καταθώσει τροπολογίες και λέω ουσιαστική προστασία δεδομένων και κάποια ελάχιστη εναρμόνιση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την πλήρη εναρμόνιση. Υπάρχει αυτή η διπλή στρατηγική και δεν ε, θεωρώ θεωρώ ότι η ελάχιστη εναρμόνιση συμβαδίζει με τα απόλυτα δικαιώματα. Τέλος πάντων, σε τελική ανάλυση πρέπει να βρούμε κάποια λογική λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις ε, των δύο επιτροπών και ξεκινώ με την κυρία Μεϊντάλ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι η Miss <laughs> Δυστυχώς η Miss δεν, μπορεί να, δεν μπορούσε να έρθει και μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρου τη και να καταθέσω κάποιες σκέψεις της uh, σκιώδους εισηγητρίας εκ μέρους της ΕΜΚΟ. Πρόεδρος, μισό λεπτό. Ε, ε, έχετε χρόνο δύο λεπτά. Ευχαριστώ λοιπόν τους αδελφούς, ιδιαίτερα Γκέπχαρτ και Φως και επίσης θα ήθελε να αποσαφηνήσω ότι την οπτική γωνία της ΣΥΜΚΟ το θέμα είναι πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα στο πλαίσιο της οδηγίας και ότι οι υποχρεώσεις για καταναλωτές και επιχείρησης δεν είναι περιβολικά επιβαρυνικές. Το κείμενο είναι αρκετά δυσδρικό θα έλεγα, έχει ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων. Στο άρθρο 3 για παράδειγμα, από την οπτική μας γωνία πρέπει να συμπεριλάβουμε την παροχή υπηρεσίας εναντί στοιχείων βάσει του GDPR. Και πρόεδρε, είναι ένα ερώτημα που θέλω να θέσω στην κυρία Γκέπερτ. Όταν λέτε ότι στον τομέα των άλλων στοιχείων, κάθε άλλου στοιχείο, κάθε άλλου δεδομένου, ε, θα θέλετε να εξαιρέσετε τα προσωπικά δεδομένα, τότε ποια είναι τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι κομμάτι του GDPR Κατά τη γνώμη μας, τα προσωπικά δεδομένα ήδη την χάνουν προστασίας βάσει του GDPR και συνεπώς δεν υπάρχουν άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να περιληφθούν υπό τον τίτλο άλλα δεδομένα. Εδώ έχουμε μια σάφια και η κυρία Μέιντελ και εγώ είμαστε υπέρ της έκθεσης του κυρίου Φως στον τομέα του όσον αφορά τον ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου και εδώ σε ένα νέο τομέα χρειαζόμαστε εναρμόνιση. Τώρα βεβαίω ξεκινάμε. Όλα αυτά είναι κοινοφανή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε 100% υπέρ των προτάσεων του εισηγητού. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Κυρία Χωσιέρ. Δεν είναι εδώ. Είναι στο δρόμο από ό,τι φαίνεται. Δεν την αντικαθιστά κάποιο, όχι. Έχετε δύο λεπτά. Δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την Βιρζίνη, αλλά σύμφωνα με την κυρία Γκέπχαρτ και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία και άλλων οριζοντίων θεμάτων όσον αφορά τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και τις επιγραμμικές συμβάσεις και ιδιαίτερα όσον αφορά τα συλλογικά μέτρα επανόρθωσης για τους καταναλωτές. Αυτό θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών το ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ψηφιακό περιεχόμενο, έχει μεγάλη σημασία οι καταναλωτέ να είναι σε θέση να απολάβουν πραγματικά των δικαιωμάτων του. Θέλω λοιπόν να ξαναδούμε αυτήν την πτυχή από εδώ και πέρα. Έχουμε κάποιε τροπολογίε επί όλων αυτών των ζητημάτων. Και προ το τέλο ε, θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των συγκεκριμένων τροπολογιών υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Στάλτον. Πρόεδρε να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές. Ε, δύσκολο το δοσχέ Για μένα πάντως το κλειδί είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται με σαφείς κανόνες όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των, περιστάσεων. Δεν θέλουμε να δώσουμε προσχήματα στις εταιρείε για να μην αποζημιώνουν ή να παγιδεύουν τους καταναλωτές. Δεν θέλουμε παραθυράκια επίσης που θα δίνει τη δυνατότητα αποζημίωσης για πολύ ακριβά μηχανήματα για ασήμαντους λόγους. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Τώρα όσον αφορά τις συμβάσεις, για μένα η ελευθερία της σύνεψης συμβάσεων, ε, ένα πράγμα που πρέπει να συμβεί είναι να μπορούν οι καταναλωτές να απολαύουν χαμηλότερων τιμών με πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Δεν βλέπω γιατί πρέπει δηλαδή να μειώσουμε, να περιορίσουμε τη διάρκεια στους 12 μήνες. Και τώρα το πραγματικό κλειδί είναι τα δεδομένα. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν ότι εδώ έχουμε ανταλλάγματα, ανταλλαγή δεδομένων με υπηρεσίες. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω τη δικαιολογία. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την επέκταση σε κάθε άλλα δεδομένα. Μου φαίνεται παράξενο που η οπτική αρχή συμφωνεί. Δεν συμφωνεί με το GDPR. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι ορισμοί δεν είναι ικανοποιητικοί και τα δεδομένα από τη στιγμή που κάποιο τα έχει στην κατοχή του μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει, να τα δώσει όποιο θέλει και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό το πράγμα, να ξανασκεφτούμε αυτέ τι προτάσει όσον αφορά ιδιαίτερα τις προτάσεις από την Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Τώρα και για τη χώρα μου, αλλά και για άλλες ε, χώρες, τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ε, να μην ε, ισοπεδωθούμε προς τα κάτω, αλλά να πάμε προς τα πάνω όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι δύσκολο το θέμα. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε περαιτέρω τους επόμενους ε, μήνες μέχρι να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Ο κ. Τζαμπάσκι δεν είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάλλας. Πρόεδρε, μιλώ εκ, εκ μέρου δύο σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω να μου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ τους εισηγητές για το έργο τους. Όπως διπιστώσαμε και χθε τους σκιώδες, ε, το θέμα δεν είναι εύκολο. Το συζητούμε εδώ και ήδη έναν χρόνο και ακόμη έχουμε τόσο ανοιχτά ζητήματα μπροστά μας. Όσο πιο πολύ υπησερχόμεθα στις λεπτομέρειες της νομοθεσίας, της ψηφιακής αγοράς, βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ ψηφιακών υπηρεσιών. Υπάρχουν τόσες πολλές που δεν διευκολύνεται το έργο μας. Το θέμα είναι πάντως η αυτοσυνέπεια και η ασφάλεια δικαίου. Θεωρώ ότι κώδικας, οι σχετικές οδηγίες και το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να συνδυάζονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο όπου και οι ορισμοί θα είναι ενιαίοι. Όσον αφορά το παιδί εφαρμογή, το συζήτησαμε εκτενέστερα τα έξυπνα αγαθά, την συμβατότητα, την περίοδο εγγύησης και το βάρος της απόδειξης. Θεωρώ ότι μια έξυπνη μηχανή καφέ να έχει απεριόριστη εγγύηση, ενώ η μια κανονική μηχανή του καφέ έχει εγγύηση μόνο για δύο χρόνια. Αυτό είναι παράλογο. Ως προς το πεδίο εφαρμογή ε, πρέπει νομίζω να ταυτίζονται τα παιδεία στη, στα δύο κείμενα. Να συνειδητοποιήσουμε επίση ότι οι δωρεάν υπηρεσίε δεν είναι πραγματικά δωρεάν. Πήραμε και την άποψη του επόπτη προστασία προσωπικών δεδομένων διαβάσαμε ξανά τον σχετικό κανονισμό, πρέπει η άποψή του να ληφθεί υπόψη για να μην έχουμε συγκρούσει με τον κώδικα. Πιστεύω ότι η συμπερίληψη των λεγόμενων άλλων δεδομένων θα οδηγήσει σε σύγχυση. Φοβάμαι ότι εκεί θα συμπεριληφθούν και προσωπικά δεδομένα. Αυτά πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογή και χαίρομαι που βλέπω ότι ο κύριο Φω συμφωνεί. Να προσαφηνήσω επίση ότι εδώ μιλάμε μόνο για προσωπικά δεδομένα μόνο όταν η χρήση απαιτεί επέκταση πέραν των βασικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. Δεν υπάρχει λόγος να συμπεριλάβουμε εδώ συμβάσεις τις οποίες υπάρχει ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις του παρόχου στην περίπτωση τερματισμού σύμβασης, θα θέλαμε να διαγραφεί αναφορά στα, κάθε άλλα δεδομένα, γιατί πιστεύουμε ότι εδώ δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο καταναλωτή. Να κρατήσουμε όμω το περιεχόμενο. Τη λέξη περιεχόμενο αποτελεί πάγια πρακτική όταν κάποιο ανεβάζει περιεχόμενο ή παράγει περιεχόμενο, συνήθω μπορεί να το πάρει πίσω ή να το διαγράψει. Αυτό είναι ελάχιστη βάση για συμβασμό. Όσον αφορά τα κριτήρια συμβατότητα, αν και φαίνεται η πλειοψηφία αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στα αντικειμενικά κριτήρια, Εμεί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι λειτουργικό αυτό ο κατάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναστροφή τη παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Φοβάμαι ότι αλλιώ ε, οι διδάξει που θα εισαγάγουμε πολύ σύντομα θα είναι παροχημένε και, θα, και δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα προχωρήσουμε τώρα με την, με δεύτερη σειρά των σχεδόν εισηγητών και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ντέντε Και δεν ξέρω, μήπως θέλει κάποιος από την ΚΟΕ να λάβει το λόγο. Η πράσινη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα μιλήσω ως ε, σκιώδη συγγήτρια και των δύο εμπλεκόμενων επιτροπών. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές ε, για τη δουλειά που έχουν κάνει και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, με αυτά τα οποία εξετάζουμε τώρα, τα στοιχεία της ε, συμβατότητας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι όσον αφορά τα κριτήρια της συμβατότητας υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Και νομίζω αυτά ε, αφορούν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή αν μπορεί κανείς ως πολιτής να γράφει ό,τι θέλει, ο κατανοητής δεν είναι εύκολο γι' αυτό να διαφωνήσει. Ε, νομίζω ότι ε, στην πρώτη πρόταση ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι τροπολογίες και θα ήθελα να επισημάνω κυρίως την τροπολογία 241 σε σχέση με την ε, διαλειτουργικότητα. Εκεί είναι πολύ σημαντικό το να διευκολύνει την ανταλλαγή των καταναλωτών ανάμεσα στους διάφορους παρόχους, δηλαδή να μην ασχολείται κανείς μόνο με το συγκεκριμένο αντικείμενο, ε, γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι επιζήμιο για τους ε, καταναλωτέ και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Και επίση πρέπει να βρούμε και κάποιου όρου σχετικά με τις αθέμητε συμβάσει να προστατεύεται ο καταναλωτή, να μην αφήνεται όλο αυτό στι διαπραγματεύσει ανάμεσα στι δύο πλευρέ, όπου οι καταναλωτέ είναι πάντα η πιο αδύναμη πλευρά. Όσον αφορά τι ε, τα μέτρα αντιμετώπισης, ε, συνήθως πρόκειται για μικροπληρωμές, περίπου 99 cent. Ε, νομίζω ότι για το ψηφιακό περιεχόμενο ε, θα έπρεπε να βρούμε κάποια λύση γιατί αλλιώς θα ήταν ένα παράλογο βάρος για τον καταναλωτή να μην μπορεί να ζητήσει πίσω τα χρήματά του επειδή είναι μικρά τα ποσά. Όσον αφορά το τέλος της, το θέμα της πάψης υπάρχει μια διαφοροποίηση από την πρόταση της Κομισιόν δηλαδή οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει κανείς πίσω τα δεδομένα του, προσωπικά ή όχι, και το κατά πόσον ο πάροχος θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα. Αυτό λένε είναι ένα άρθρο στην πρόταση Κομισιόν, αλλά δεν είναι πάντα το ίδιο, γιατί αν μιλάμε για ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο συνδημιουργείται από τους χρήστες της πλατφόρμας, βεβαίως και θα πρέπει ο χρήστης να κατεβάζει αυτό το περιεχόμενο, αλλά δεν θα πρέπει και ο πάροχος ε, να διαγράφει το περιεχόμενο της ε, πλατφόρμας. Εγώ λοιπόν προτείνω ε, να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Όσον αφορά το θέμα των δεδομένων ως ε, ανταπόδοση. Ε, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την πρόταση των καταναλωτών, αλλά να βρούμε και κάποια λύση η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ε, βρούμε κάποια λύση. Όσον αφορά τους όρους των συμβάσεων, εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι καλύτερα να υπάρχουν μακροχρόνιες συμβάσεις, γιατί ξέρετε είναι κυρίως ο ανταγωνισμός ο οποίος είναι καθοριστικός. Γι' αυτό εγώ προτείνω να περιορίσουμε χρονικά τις ε, συμβάσεις. Και επ' αυτού θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτή την πρόταση και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κώδικα επικοινωνίας. Γιατί ορισμένες υπηρεσίες επικοινωνίας που είχαν προβλεφθεί αρχικά ε, με πιο ε, βραχύβιες συμβάσεις τώρα πλέον περιλαμβάνονται στην οδηγία που προβλέπει μεγαλύτερες χρονικές χρονικές περιόδους. Ε, θέλω, επιθυμώ οι δύο αυτές προτάσει να συμβαδίζουν και να μην αντιβαίνει ή να μην αντίκειται η μία στην άλλη. Grazie. Ringrazio anch'io i correlatori perché hanno un compito eh, veramente... Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συζητητές γιατί έχουν πολύ δύσκολη δουλειά. Κοιτάξτε, εκείνο που δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτή την έκθεση είναι ε, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ε, σιγουριά του δικαιώματο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλέ οδηγίε ε, που αφορούν σε θέματα ψηφιακά, έχουν σχέση και με τα προσωπικά δεδομένα και με τον κώδικα των τηλεπικοινωνιών. Εγώ πιστεύω ότι οι τιμές μέγιστη προσπάθειά μας θα πρέπει να την αφιερώσουμε στο να υπάρχει ένα αρμονικό πλαίσιο. Να μην υπάρχουν επικαλύψεις γιατί αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικούς νομικούς ορισμούς ε, και να δυσχεράνει το έργο μας. Εγώ λοιπόν επιθυμώ να υπάρχει μια προσαρμογή ε, στους κανόνες όσον αφορά τις επιγραμμικές πωλήσει. Τώρα θα μπω λιγάκι στην ουσία του θέματος. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ευχαριστημένος με τις διευκρινήσεις που έδωσαν οι συγητές γιατί αυτή η οδηγία δεν αντικαθιστά επουδενή την οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό καταρχήν ως σημείο αφετηρίας. Κατόπιν, όσον αφορά το περιεχόμενο υπηρεσιών, ψηφιακών υπηρεσιών, νομίζω ότι εδώ πρέπει να ορίσουμε ένα σαφέστερο πλαίσιο προστασίας για τους καταναλωτές και θα ήθελα να κλείσω με μια παρατήρηση που θέλω να κάνω σχετικά με το περίφημο embedded software όπως αναφέρθηκε και συζητήθηκε και χτες. Οι συγητές ε, προτείνουν μια λύση που αφορά στο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο θα εντάσσεται, θα συμπεριλαμβάνεται ε, σε κάποιες ε, ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εγώ θεωρώ ότι η προστασία του καταναλωτή σημαίνει να υπάρχει σαφήνεια. Και η, ο πιο ε, σύντομος ορισμός είναι αυτός που προτείναμε χθε. δηλαδή να μιλάμε μόνο για περιεχόμενο προεγκατεστημένο. Αυτό είναι μια ε, σαφέστερη προσέγγιση που νομίζω ότι διευκρινίζει κατά κάποιον τρόπο το τι πρέπει να κάνουμε. Thank you very much. Ε, Madame ENF. Ευχαριστώ, ENF. Ε, κάποιος άλλος από το ΕΝΕΦ, e όχι. Δεύτερος γύρος τότε, των σχεδόν εισηγητών. Μήπως κάποιος άλλος επιθυμεί το λόγο. Αν όχι, νομίζω έχουμε ακόμα χρόνο να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Έτσι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και θα εστιάσω στα ζητήματα που έθιξαν διάφοροι ομιλητές για τα, προσωπικά δεδομένα. Χαιρόμαστε που θεωρούν οι επιτροπέ σα ότι πρέπει να περιληφθούν εδώ στο πεδίο εφαρμογή. Αυτό είναι σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε όμως ότι θα υπάρχει αντίρρηση για το GPDR όσον αφορά του στόχους, για να μην υπάρχουν δηλαδή αντιφάσεις εκεί. Και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη η έκθεση του εποπτικού οργάνου, του ευρωπαϊκού, που είναι ενδιαφέρον ότι υποστηρίζει, όπως αναφέρει και παραθέτω, το στόχο για την ενίσχυση, για την προστασία των καταναλωτών, από τις οποίες απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο σημείο της έκθεσης αυτής, γιατί αυτό που κάνουμε με την πρόταση δημιουργούμε επιπρόσθετη προστασία για τους καταναλωτές ως καταναλωτές αυτούς καθεαυτούς πέραν δηλαδή του περιεχομένου και αυτό είναι ο στόχος της πρότασης ο κ. Τόλτον είπε ας πούμε ότι η γνωμοδότηση του DDPS ε, δεν θα πρέπει τα δεδομένα να οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα κτλ. Όντω αυτό λέει το DDPS. Και όπως και η κυρία Ρέιντα, θεωρώ και εγώ ότι μπορούμε να βρούμε μια σχετικά εύκολη λύση. Και έχει κάνει προτάσει και του EDPS επ' αυτού. Να ευκαιρίσουμε λέει το πεδίο εφαρμογής αλλά να παραμένουν τα προσωπικά δεδομένα στο πεδίο εφαρμογή. Δεύτερο, τα λοιπά δεδομένα. Και εκεί πέρα έχει νομίζω δίκαιο. Ένας από τους λόγους για την περίληψη των λοιπών δεδομένων είναι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα προσωπικά δεδομένα, περίπλοκος ορισμός και υπόκειται βεβαίω και στην ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τα λοιπά, τα υπόλοιπα δεδομένα. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε να απελευθούν και τα δύο, και τα προσωπικά και τα λοιπά δεδομένα στο πεδίο ώστε να μην βαρύνουμε την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας με ενδεχόμενα προβλήματα προσδιορισμού. Βεβαίω έχουμε και οικονομική αξία στα δεδομένα. Λάβετε υπόψη, ας πούμε, παραδείγματι τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εσάς ως κατανοτές. Ας πούμε, σας αρέσει τα ταινία. Ή, ξέρω εγώ, άρενε θεατέ, ηλικία 32 με 50, οι οποίοι τέλο πάντων παρακολουθούν κάποιε σειρέ κτλ. Αυτό το κάνουν ας πούμε, στο Netflix και η σειρά πούμε, House of Cards ε, σε αυτό βασίστηκε. Υπάρχει λοιπόν οικονομική αξία εδώ και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προστατευτεί, να συγγνώμη, περιληφθεί στην πρόταση. Και το εποπτικό όργανο επίσης αναγνωρίζει ότι θα είναι πιο προσωπαγή τα δεδομένα μελλοντικά. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε ε, βεβαίως ανώνυμα δεδομένα και θα πρέπει να λάβουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Το λέω αυτό επειδή επίσης η Κομισιόν αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της εφαρμογής. Έχουμε ξεκινήσει και μια μελέτη συγκριτική για όλους τους χώρου μέλη για το πώς εφαρμόζονται οι για το collective address όλες τις χώρες μέλη. Ένα θέμα νομίζω οριζόντιο και νομίζω δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε με δύο λόγια μόνο σε αυτή την πρόταση και είναι σημαντικό νομίζω η Κομισιόνα να του δώσει την ιδιαίτερη σημασία για αυτό που λέμε collective address. Και τέλος, ένα τελευταίο σημείο. Ο κώδικας ηλεκτρονικών ε, τηλεπικοινωνιών αναφέρθηκε από διάφορου βουλευτέ και συμφωνούμε. Θέλουμε και εμείς να υπάρχει μια συνεπή πρόταση. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο και εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε τον ορισμό όπως είχε προηγουμένω. και που τώρα βρίσκεται δηλαδή στις ηλεκτρονικές ε, τηλεπικοινωνίε. Για δύο λόγους. Καταρχάς η πρόταση έχει μια γενική φύση, δηλαδή όπου υπάρχουν επιμέρους ζητήματα να ρυθμίζονται στις επιμερούς διατάξεις. Αυτό αφορά τις οικονομικές υπηρεσίε, την υγεία και πολλά άλλα θέματα. Και θέλουμε να παραμείνουμε στην πρόταση αυτή και να αφήσουμε τα επιμέρους ζητήματα στους ειδικού. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει μια ισοτιμία. Στις τέσσερις κατηγορίες των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή ανεξάρτητη πάροχη κτλ. που περιλαμβάνονται στην οδηγία, και εκεί θα θέλαμε να υπάρχει μια ισοτιμία. Δηλαδή, πάροχη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και λοιπόν Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτά που κάνουμε, να υπάρχει αυτή η ισοτιμία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να ξαναδώσω τώρα το λόγο στους συνεισηγητές Ποιος θα ήθελε το λόγο πρώτος. Η κυρία Γκέπχαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Σουβάμπ. Την ερώτηση που μου την έκανε πολύ νωρίς σήμερα το πρωί και με ρώτησε τι εννοώ όταν μιλάω για δεδομένα που δεν σχετίζονται με άτομα, αλλά είναι κάποια άλλη μορφή. Εγώ επισκέφθηκα στη Λίλ ένα, μια εταιρεία για την κυβερνοασφάλεια και εκεί μου επισήμαναν το πόσο σημαντικό είναι να συμπεριληφθεί αυτή η διευκρίνηση. Και ένας άνθρωπος που δουλεύει εκεί μου είπε ότι είναι τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών apps. Αυτά αποθηκεύονται μεμονωμένα και ε, με τη διασύνδεση τώρα των ε, δεδομένων ε, επαναφέρονται και αφορούν άτομα. Να σας πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω το δικό σας το τηλέφωνο, αλλά εγώ στο δικό μου το iPhone, έχω iPhone, λοιπόν στο iPhone μου έχω το WhatsApp, το οποίο WhatsApp μπαίνει στις επαφές μου και έχω και τα Google Maps, τα οποία τα χρησιμοποιώ για να πάω κάπου. Αυτά τα δύο δημιουργούν δεδομένα που έχουν σχέση με άτομα. Και όταν τώρα βάζω μία διεύθυνση στα Google Maps, ε, γιατί κάπου θέλω να πάω, και αυτό συνδυάζεται με ένα άτομο το οποίο έχω στις επαφές μου, αυτομάτως δημιουργούνται νέα δεδομένα τα οποία έχουν σχέση με άτομα. Δηλαδή τι φαίνεται, α, η κυρία Γκέπχατ πάει να επισκεφτεί τον τάδε στο τάδε μέρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να καλύπτονται και με τον ορισμό ε, τον οποίο έχουμε για τα δεδομένα που δεν αφορούν άτομα δεν καλύπτονται όμως. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με τον κύριο Steinmeier ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομική ασάφεια και ανασφάλεια. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτά τα any other data για να μην αρχίσει οποιαδήποτε νομική αντιπαράθεση. Εγώ δεν θέλω να δίνω δουλειά στους δικηγόρους. Αυτοί δηλαδή να λένε τι είναι δεδομένα ε, μη προσωπικής φύσεως. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ε, δημιουργούμε νομική ε, ασφάλεια. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Και το άλλο, τα δεδομένα όσα ανταπόδοση, όπως το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Διότι αυτά τα δεδομένα τα αποκαλούμενα δωρεάν apps, αυτά τα παιχνίδια και όλα τα άλλα τα οποία μπορεί κανείς να τα ανεβάσει δωρεάν, αυτά είναι παιχνίδια τα οποία προσφέρονται. Εγώ ξέρετε έχω δει και apps που προσφέρουν και υπηρεσία αφύπνισης, παρότι κάθε τηλέφωνο έχει ξυπνητήρι, δεν το χρειάζεται αυτό ε, κανείς. Το προσφέρουν όμως οι υπηρεσίες, ξέρετε γιατί, για να βάλουν χέρι στα δεδομένα. Και γι' αυτό λοιπόν ε, είναι ιδιαίτερα προβληματικό το ότι δεν αναγνωρίζονται αυτές ε, οι αντιπαροχές. Εγώ ειλικρινά είμαι κατά της εμπορευματοποίησης των δεδομένων, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα και ως εκ τούτου θεωρώ, και εδώ δίνω απόλυτα δίκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα δεδομένα ως ανταπόδοση θα πρέπει να τα κρατήσουμε έτσι ώστε η προστασία που προσφέρεται να διευκρινίζεται και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι πράγματι κάναμε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τους κινδύνους και έχω και μία ερώτηση και εγώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, άκουσα από εσάς ότι ε, συλλογικές αποζημιώσεις δεν πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στο κείμενο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει έχει κάποιες επιφυλάξεις επί του θέματος και θέλω πραγματικά να γνωρίζω πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείτο, αρνείτο κατηγορηματικά να επεξεργαστεί μια πρόταση και να την καταθέσει στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, να μην μας ξεφορτωθείτε με κάτι που δεν προτίθεστε να κάνετε, να μας διαβεβαιώσετε για κάτι που πραγματικά έχετε πρόθεση να επιβάλλετε. Ο κύριος Φώστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα ε, όσον αφορά τα ε, θέματα που έχουν σχέση με άτομα, να επανέλθω λιγάκι σε αυτό το θέμα. Βεβαίω είναι αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε έναν εντεταλμένο για δεδομένα θα μας πει αυτό που ακούστηκε προηγουμένως. Όμως δεν είναι αυτή η όλη έννοια του εγχειρήματο για τους ε, εντεταλμένους ε, για δεδομένα. Η χρήση ενός ε, κινητού αυτή και μόνο είναι επικίνδυνη γιατί εκεί αυτομάτως προκύπτουν δεδομένα. Τι θέλω να πω, να τα δούμε λιγάκι σχετικά τα πράγματα. όσον αφορά αυτή την τοποθέτηση συμφωνώ αλλά δεν πρέπει κανείς να θεωρεί ότι το EDPS είναι νομοθέτης. Νομοθέτης είμαστε εμείς και δεν θα πρέπει να το ε, αμφισβητούμε. Καλά, καλό αυτό που ελέγχθη, αλλά σας είπα και κάποιες επιφυλάξεις. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό δεδομένων που αφορούν άτομα και άλλη μορφής δεδομένα. Αν θυμάμαι καλά, στην βασική ε, οδηγία, θεμελιώδη οδηγία για την προστασία των δεδομένων, ορίζουμε ποια είναι τα άλλη φύσεως δεδομένα. Αυτά που δεν έχουν σχέση με άτομα δεν συμπεριλαμβάνονται. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στην εξή δυσκολία. Στον ορισμό μας θα πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι άλλη φύσεως δεδομένα. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν στο τέλος να διαγράφουμε ή να δίδουμε πίσω τα άλλη φύσεω δεδομένα. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Κανείς ε, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποια δεδομένα ανήκουν σε ποιον αν κάποιος ας πούμε ε, ολοκληρώσει μια σύμβαση και ζητήσει από τον εργοδότη ε, να του βρει στα δεδομένα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί δεν ξέρει ποια είναι προσωπικά και ποια όχι. Άρα δηλαδή προκύπτει πρακτικής ε, φύσεως ε, πρόβλημα. Το τι πρέπει να κάνουμε με αυτά τα any other data. Από πλευρά ορισμού το μόνο που μπορεί να ισχύσει είναι ότι τα any other data περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και ο ορισμός είναι ε, ο εξής, ε, το να συνδυάζονται κάποια δεδομένα και να αφορούν ένα άτομο, έναν άνθρωπο, αυτομάτως είναι δεδομένα τα οποία ε, κατά την άποψή μου προστατεύονται. Για μένα, αυτά τα any other data δεν χρειάζεται να τα συμπεριλάβουμε και ακόμα και αν συμπεριληφθούν θα πρέπει να διευκρινιστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην αποτελούν ιδιαίτερη επιβάρυνση καταρχήν για να οριστούν. Και αυτό είναι κατά της αρχής της προστασίας δεδομένων, ότι δηλαδή καταρχήν εντοπίζονται τα δεδομένα για να μπορούν μετά να διαγραφούν. Δεν είναι αυτή η ουσία του όλου θέματος. Τώρα, όσον αφορά στη νομική ασφάλεια, ε, συμφωνώ απόλυτα. Πράγματι, χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια και ε, εδώ πρόκειται για την οδηγία e-Privacy Directive Communication Code. Σε όλα αυτά ε, χρειαζόμαστε ε, λογικούς ε, ορισμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα λογικό πλαίσιο να έχουμε ένα σχέδιο. Αυτή τη στιγμή ε, τυχαία βαδίζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, ποιος κάνει τι ε, και νομίζω ότι ο διαχωρισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος γιατί υπάρχουν μοντέλα τα οποία καλύπτονται από διάφορες οδηγίες αλλά επειδή δημιουργούμε όλα αυτά τα εμπόδια ενδεχομένως τελικά να μην γίνει τίποτα, να καταλήξουμε σε αδιέξοδο. Ως εκ τούτου εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όσον αφορά τώρα τις ε, μακροχρόνιες ε, συμβάσεις, ένα θέμα που ετύγει. Με συγχωρείτε, έχει την καλωσία να τελειώνετε. Ε, τελείωσα. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Στάντμαια, θέλετε εσείς ε, να απαντήσετε σύντομα στην ερώτηση της κυρίας Γκέπχαρτ. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Εμείς λαμβάνουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά, το collective address Έχουμε συστάσεις για το πεδίο εφαρμογή και θα πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει, τι έχουν εφαρμόσει οι χώρες μέλη. Από πρώτα στοιχεία έχουμε μια εικόνα, αλλά όχι πλήρη. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάποιους ελέγχους, κάποιες επαληθεύσεις πριν αποφασίσουμε. Πάντως, σας διαβεβαιώ, το λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά. Να δούμε την υπόθεση Volkswagen. και τις προσωπικές προσπάθειες της Επιτροπής σας διαβεβαιώ το λαμβάνουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά. Και να πω στον κύριο Φως ότι συμφωνώ απόλυτα για τα άλλη φύση δεδομένα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τη φύση τους. Και εκεί όπου χρειαστεί θα δείξουμε ευελιξία, ώστε να βρούμε δηλαδή ώστε να έχουμε μια έτσι, τελική μορφή κειμένου που θα λαμβάνει υπόψη αυτά που ο κύριος Φως. ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος της κοινή συνεδρίασής μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Χαρενσέσο Βάφο για την συμπροεδρία και θα ήθελα να σας καλέσω να κατεβούμε τώρα κάτω στον τρίτο στην είσοδο της Ολομέλειας για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομακαρικής ενέργειας της Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ θα ήθελα να σας επιθυμίσω στα μέλη της ομάδας μας ότι θα ξεκινήσουμε στις 10 και 4 στο 5G3, στην 5G3. Ευχαριστώ πολύ.